Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre réunion, la première de l'année, hein, je crois. Oui. Euh, Ως ε, πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, έχω την τιμή να προεδρεύσω στην ε, συνάντησή μας για τη Μέση Φουτία την συνεδρίαση καταστατική συνεδρίαση. Θα προεδρεύσω λοιπόν προσωρινά μέχρι να εκλεγεί ο ή πρόεδρός μας. Ε, κυρίσω την έναρξη τη συνεδρίαση και θυμίζω το στόχο τη συνάντησή μα να, να εκλέξουμε το Προεδρείο της ε, Επιτροπής πρώτον τον πρόεδρο και μετά έναν έω τέσσερι αντιπροέδρου βάσει του άρθρου 191 του κανονισμού. Θα πρέπει πρώτα να εκλέξουμε τον ή την πρόεδρο και μετά του ή τι αντιπροέδρου. Για να διεξαχθεί σωστά η ψηφοφορία θα πρέπει σε πρώτη φάση και πριν οργανωθεί η ψηφοφορία να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν και αναπληρωτέ ή μόνιμοι αναπληρωτέ και σα θυμίζω ότι βάσει του άρθρου 187 το όνομα των αναπληρωτών που δεν είναι μόνιμοι θα πρέπει να μου έχει κοινοποιηθεί πριν την ψηφοφορία. Έχουμε τον κύριο Τσάμπα Ορή, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Φιλίπ Κασμάρεκ. Είστε παρόν κύριε πριν λοιπόν την ε, ψηφοφορία αυτή καθεαυτή, θα ήθελα να προχωρήσουμε σε δύο προηγούμενε διαδικασίε. Πρώτα απ' όλα να επαληθεύσουμε ότι υπάρχει απαρτία. Ναι, βάσει το άρθρο 195. Εν, μια απαρτία σε από 8 μέλη. Και τώρα θα δούμε τι υποψηφιότητε υπάρχουν για την Προεδρία τη Επιτροπή. Υπάρχουν υποψήφοι για την Προεδρία, κυρία Γκρέζ. Εάν μου επιτρέπετε, αφού έχω την τιμή ως συντονίστρια της ομάδας των προσύνων, να σας υποβάλω την υποψηφιότητα της κυρίας Εύα Ζολή για να αναλάβει την Προεδρία αυτή τη επιτροπή. Si Donc, est-ce que le candidat émane d'un groupe politique moins 5% Εάν υπάρχει παρουσία 5% των ε, πλήρων μελών, ναι, είναι η απάντηση. Επίσης, εάν συμφωνούν οι υποψήφοι, ναι. Δεν χρειάζεται νομίζω να το ρωτήσω. Όχι, πρέπει να ρωτήσω την κυρία Ζολή. Κυρία Ζολή, δέχομαι με ιδιαίτερη ευτυχία αυτήν την ε, αποστολή. Η υποψήφια έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών σφαιρόντων. Ναι. Ωραία λοιπόν. Θα έλεγα να ψηφίσουμε διαβοή. Ναι. Voilà. Donc, euh, ce vote a été fait. Ωραία λοιπόν, εκλογή διαβοήση. Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα του ή άλλω. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχεί που η κυρία Ζολή θα συνεχίσει και στο υπόλοιπο της θητείας στην Προεδρία της. Κυρίσουμε λοιπόν, βάζει το 191 εδάφιο πρώτο, πρώτη παράγραφος εδάφιο δεύτερο, την εκλογή της κυρίας Ζολή διαβοής. Θα ήθελα να σας εκφράσω, κυρία Ζολή, την χαρά μας που μπορείτε να συνεχίσετε τη δραστηριότητά σας ως πρόεδρος της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας καλέσω να αναλάβετε εσείς το φακό της Προεδρίας ως πρόεδρος της Επιτροπής στο Προεδρείο. Ευχαριστώ merci. Je την κυρία Στιφλέρ που δέχτηκε να αναλάβει την διεξαγωγή αυτής της ψηφοφορίας και που τα έκανε τόσο αποτελεσματικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχηθώ κάθε ευτυχία για το 2012. Όσους δεν είχα την τύχη να τους συναντήσω, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο κυρίως. Επίσης, θέλω να σας, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά που μου αναθέσατε την εμπιστοσύνη σας. Όταν ξεκινήσαμε τη θητεία αυτή το 2009, υπέστημε τις πρώτες συνέπειες της ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Προτεραιότητά μας τότε ήταν να προασπίσουμε τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και την αναπτυξιακή πολιτική για την ανάπτυξη και τη βοήθεια για την ανάπτυξη, παρόλο που ήταν πολλέ οι χώρε που αποφάσισαν να μειώσουν ε, τα κονδύλια που απευθύνονται στην αναπτυξιακή βοήθεια. Τώρα η κρίση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, χτυπώντας ξεχωριστά τα διάφορα κρατημέλη και κάποιοι πλήττονται ιδιαιτέρως. Έχουμε εδώ το το καθήκον να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις συνέπειες του καθημερινού βιώτων των πολιτών και να ξαναδώσουμε ελπίδα και πίστη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να μην ξεχνάμε ωστόσο ότι οι χώρες του Νότου επίσης ε, υποφέρουν από τις συνέπειες της κρίσης πέραν των ε, καταστροφικών συνεπειών των κλιματικών αλλαγών. Έτσι λοιπόν ε, το καθήκον μας θα είναι ακόμη πιο δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει μάλλον να σα εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι θα με στηρίξετε σε όλε αυτέ τι προσπάθειε γιατί γνωρίζω την αγωνιστικότητά σα και την αποτελεσματικότητά σα. Χάρη σε αυτέ τι προσπάθειε, έχουμε αναλάβει κάποιε φορέ το ρόλο ενό απλού συμβούλου, ενώ μα έχουν εμπιστευτεί με την ψήφο του τόσα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε για να λάβουμε ένα ρόλο πιο δραστικό. Σα ευχαριστώ λοιπόν εκ νέου για την εμπιστοσύνη σα και σα καλό να συνεχίσουμε την ψηφοφορία για να εκλεγεί το Προεδρείο της Επιτροπής μας. Προχωρούμε λοιπόν στην εκλογή των τεσσάρων αντιπροέδρων ανδρών γυναικών, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Θα ήθελα να δούμε τι υποψηφιότητες υπάρχουν για τη θέση της πρώτης αντιπροέδρου ή του πρώτου αντιπροέδρου. Θα ήθελα να προτείνω ως πρώτη αντιπρόεδρο την κυρία Στρίφλερ, ως δεύτερα τον κύριο Ντέβα και ως τρίτο την κυρία Τσανική. Ευχαριστώ. Άλλη υποψήφια, κύριε Μαρτίνεφ. Μικρό. Το μικρόφωνο σα, λέει ο πρόεδρο. Voilà, merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σα. Socialistes, nous voulons présenter la candidature de Madame Κρέτσου. Je ne sais pas si c'est pour... Κυρία Κρέτσου, για την πρώτη αντιπροεδρία ή για τη δεύτερη προτείνεται από εμά του σοσιαλιστάς και έχει αφήσει εδώ ένα χαρτάκι για να βεβαιώσει ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα. Δεν ξέρω όμω ε, ε, αν πρόκειται γιατί τη θέση της πρώτης αντιπροέδρου ή τέταρτη. Απλώς το σας το λέω για να το λάβετε υπόψη. Πώς το γιατί θέσετε την πρόεδρο, οπότε τώρα θα μείνουμε για τις προσθέτες για την πρώτη αντιπρόεδρο ή τον πρώτο αντιπρόεδρο. D'accord. Monsieur Newton Dunn, vous avez la parole. Κύριε το λόγο. Δεν με έχετε μπερδέψει. Εγώ θέλω να πω είναι η ψηφιότητα Ντέβα, δεύτερη ψηφιότητα. Μεγάλη μα τύχη να συμμετέχει εδώ, γιατί ήταν προ του Κοινοβουλίου. σχεδόν εκτό από με κάποιε εκατοντάδε ψήφου ε, για κάποιο θέμα. Καθαρά τεχνικό δεν ε, διαδικαστικό δεν επανεξελίχθηκε. Εγώ τον προτείνω για αντιπρόεδρο τη Επιτροπή μα, όχι, όχι, όχι, να τελειώσουμε με την πρώτη αντιπροεδρία, λέει η ε, Δεν έχουμε άλλες υποσχέσεις για τη θέση αυτή. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει τώρα να ε, ζητηθεί είναι ε, για τη Μουσική Στίφλερ ε, κατά πόσον ε, δίνεται, κυρία ε, από πολιτική ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, από 25% ή 5%. Η απάντηση είναι ναι. Κυρία Στίφλερ, εσείς ε, συμφωνείτε ε, για την υποσχετά σας να είστε η πρώτη μας ε, αντιπρόεδρος. Ναι, ναι. μεγάλη χαρά κύριε Ζωηλή, σας ευχαριστώ. Συμπληρώσατε την δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα όπως προβλέπει το πρώτο παράρτημα. Ναι, ναι. Οκ, okay. και τότε σας προτείνω μια που δεν έχουμε ε, άλλους για την θεσία αυτή. Με τον κυρία Στίφνη σας προτείνω ψήφο με ε, διαβοής. Επομένως, διαβοής η Στίφνη θα εξελέγει σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 2. Πρώτο εδάφιο. Σας ευχαριστώ κύριε Στίφλερ και τώρα θα προβούμε στην εκλογή ε, του συναδελφού ή τη συναδελφού για τη θέση του Δευτερού Προέδρου και τώρα να δούμε ποιε είναι οι υποψηφιότητε για τη δεύτερη υποψηφιότητα. Αυτή είναι για το δεύτερο αντιπρόεδρο. Προτείνω όπω και προηγουμένω τον κύριο Στυμπά. Est-ce qu'il y a d'autres candidats Υπάρχουν άλλε υποψηφιότητε για τη θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου ή δευτέρας αντιπρόεδρου. Στηρίζεται από μια πολιτική ομάδα η δευτερου αντιπροεδρου στηριζεται απο αυτή από το 5% των μόνιμων μελών βάσει του άρθρου 13.1. Η απάντηση είναι ναι. Κύριε Ντέβα, θέλετε να γίνετε ο δεύτερος αντιπρόεδρός μας. Έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεβά. Έχετε συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικού ενδιαφέροντος όπως προβλέπετε στο παράρτημα 1 του κανονισμού. Πολύ ωραία. Εφόσον δεν υπάρχουν τις υποψηφιότητε για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου, ορίζουμε τον κύριο Ντέβα διαβοή. Ο κύριος Ντέβα είναι εκλεγμένος διαβοής βάσει του άρθρου 191 παράγραφος 2 του κανονισμού μας. Τώρα να περάσουμε στην εκλογή του τρίτου αντιπρόεδρου ή της τρίτης αντιπρόεδρου. Υποψήφοι για την θέση του τρίτου ή της τρίτης αντιπρόεδρου. Πρώτα η της τριτης αντιπροεδρου εκεί. <coughs> Merci beaucoup. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Άλλοι ή άλλες υποψήφοι για τη θέση της τρίτης ή του τρίτου αντιπρόεδρου. Η πρόταση αυτή στηρίζεται από πολιτική ομάδα. Η κυρία Τζανίκη έχει δώσει τη γραπτή της συγκατάθεση για την υποψηφιότητα αυτή και έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικού συμφέροντος. Μπορούμε λοιπόν να εκλέξουμε την κυρία Τζανίκη διαβοής. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει εκλεγεί η κυρία Τζανίκη διαβοής. Και τώρα, πριν την ψηφοφορία υποψηφιότητα για τη θέση του τετάρτου ή της τετάρτης αντιπρόεδρου. Κύριε Μαρτίνεφ. Um, euh, euh, κυρία Πρόεδρε, θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν από λίγο. Εγώ προτείνω την κυρία Κρέτσου, την κυρία Κορίνα Κρέτσου για τη θέση αυτή. Νομίζω ότι έχει υποβάλει τη συγκατάθεση της γραπτός και επίσης τη γραπτή βεβαίωση ότι έχει υποβάλει την ε, δήλωση οικονομικού συμφέροντος. Ναι, η ομάδα αυτή λοιπόν στηρίζεται από μια πολιτική ομάδα και στηρίζεται τουλάχιστον από το 5% των ε, τακτικών μελών της Επιτροπής. Υπάρχει γραπτή συγκατάθεση της κυρίας Κρετσού και έχει συμπληρωθεί και η δηλώση οικονομικού συμφέροντος από την ενδιαφερόμενη. Προτείνω λοιπόν διαβοής να εκλέξουμε την κυρία Κρετσού. je déclare κυρία του έχει εκλεγεί διαβοής. Euh, Καλό τώρα τους και τις αντιπροεδρούς που επανεξελέγησαν και βρίσκονται στην αίθουσα και τους οποίους πρέπει να συγχαρώ βεβαίως θερμά να έρθουν στο Προεδρείο και να αναλάβουν τις θέσεις τους στο πλάι μου.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 και τώρα περνάμε στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, διάφορα εφόσον υπάρχουν. Δάλλως κηρύσουμε τη λήξη της καταστατικής συνεδρίασης. Έχετε ενδεχομένως διαδικαστικά σημεία τα οποία θα θέλετε να συζητήσουμε. Εγώ από την πλευρά μου δεν έχω κάτι. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους για τη συμμετοχή σας στην καταστατική μας συνεδρίαση και σας δίνω ραντεβού αύριο το απόγευμα για την τακτική μας συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε, θα έχουμε την τύχη να υποδεχτούμε και πάλι τον κύριο Bill Gates. Σας θυμίζω ότι ξεκινάμε στις 2 το απόγευμα και όχι στις 3. Και θα συναντηθούμε στο ημικύκλιο. Κυρίσω την λήξη της καταστατικής συνεδρίασης. Merci.